Good evening, colleagues, ladies and gentlemen. Γεια σας κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο κύριος Μπούζεκ. Τι να σου πω, περπάταγα 10 λεπτά από το κτίριο Τουρ στο 11-12 για να έρθω εδώ σε αυτήν την συνεδρίασή μας της Επιτροπής. Αλλά ευτυχώς το σημαντικό το καταφέραμε να έχουμε κοντά μας την εισηγήτρια. Για να Έχουμε το σχέδιο μέσα διάταξη για σήμερα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχουμε ένα, ένα θεματάκι μόνο. Συμφωνείτε, συμφωνείτε από ό,τι βλέπω και επιτρέψτε μου να σας πω από το τρίτο. Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Και έχουμε επίσης το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού 1 2015 για το ΕΦΣΥ, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων. Οπότε θα πρέπει να συζητήσουμε το σχέδιο νομοδότησης. Επίσης, πρέπει να ευχαριστήσω την ε, κυρία Συγήτρια και τους σκιώδης εισηγητάς, διότι τα κατάφεραν. Ετοίμασαν το σχέδιο κειμένο μέσα σε όλη αυτή τη δουλειά που είχαν, γιατί επίσης έμαθα ότι με τους σκιώδης εισηγητές η εισηγήτρια συναντήθηκε πολλές φορές. Μόνο στα αγγλικά όμως έχουμε το σχέδιο της γνωμοδότησης. Για κοιτάξτε και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Και λέει ότι ζητήθηκε από τις μεταρρυθμιστικές υπηρεσίες να το έχουν έτοιμο το κείμενο εγκαίρως για την κατάδυση των τροπολογιών, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. In all the languages. So we should expect all the amendments additional because... Οπότε, μπορείτε να δείτε στο σχέδιο κειμένου τέλο πάντων ποιε είναι οι υποβληθήσει ε, τροπολογίε μέχρι τώρα. Όλες, όλες θα μεταφραστούν. Let me remind you. Και σας υπενθυμίζω. Δε. Δυνάμει του άρθρου 54 του οργανισμού έχει αποκλειστική αρμοδιότητα η Ήτρε. Και για τους στόχους του άρθρου 5 πράγματος 2 όπως προβλέπεται για το ταμείο αυτό το ΕΦΣΙ και επίσης ε, σύμφωνα με το 18 και το 20 τα άρθρα όσον αφορά τις ε, περικοπές του ορίζον 2020 και του Κοινωνικού Ταμείου. Οπότε θα πρέπει να δούμε τώρα Οπότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το ταμείο αυτό, όσον αφορά τον προπολογισμό του. Και ευθύ αμέσω για πέντε λεπτά θα δώσουμε στην κυρία Φανμπρίντ το λόγο. Πέντε λεπτά σας αρκούν. Καλά, άντε έξω. Um, θα κάνω ό,τι μπορώ, κύριε μου. Ήδη έχουμε εμπειρία να κινούμαστε πολύ γρήγορα για αυτό το θέμα. Είχαμε πολύ λίγο χρόνο για να γραφτεί η έκθεση Ξέρω ότι υπάρχει λίγος χρόνος και για τη σύνταξη των τροπολογιών, περιορισμένος χρόνος επίσης για τη σύνταξη συμβιβαστικών και να φτάσουμε μετά πάλι γρήγορα μέχρι τη ψηφοφορία και τη διαβούλευση με το Συμβούλιο. Συνεργαστήκαμε όμως καλά με τους κοιόδης, τα υπόλοιπα μέλη καθώς και εκτός κοινοβουλίου ανθρώπους για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια άποψη πιο συγκεκριμένη. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα μέλη της γραμματείας μας που εργάστηκαν πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά αλλά και από άλλες γραμματείες πολιτικών ομάδων αρχίζω επαναλαμβάνοντας κάτι η έκθεση περιλαμβάνει επικρίσεις αλλά αυτό όχι γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο αυτό το εύση που λένε την κύρια ιδέα του την υποστηρίζουμε πρέπει να υπάρξει πρωτοβουλία για στρατηγικές επενδύσεις και επιτέλους η Κομισιόν φαίνεται να μετακινείται από την πεποίθησή της ότι μόνο η λιτότητα αξίζει τον κόπο. Έτσι είναι απαραίτητη η συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών μεταξύ άλλων για να δημιουργηθεί μια καινούργια Ευρώπη. Θα ήθελα επίσης να τονίσω γενικότερα ότι τα τελευταία δύο χρόνια Ακούστηκαν προτάσεις για προγράμματα κοινωνικής συμπερίληψης, κλιματολογικών αλλαγών, ενεργειακή ανεξοικονομήσεων κλπ. Και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το ΕΦΣΙ αυτό θα ευθυγραμμίζεται όχι μόνο με αυτά τα προγράμματα και τις προτάσεις, αλλά θα αποτελέσει και το όργανο που θα μπορέσει να τις πραγματοποιήσει αυτές τις ιδέες. Και αυτό μέσω της στήριξης επενδύσεων στους στρατηγικούς τομείς που να καταλήγουν σε μια βιώσιμη οικονομία χωρίς πολλά διοξίδια με περισσότερες ανανεώσιμες πηγές, με την ψηφιακή οικονομία και φυσικά με την έρευνα και την καινοτομία. Τώρα συγκεκριμένα στοιχεία της έκθεσης. Είχα πει ότι θα τονίσω ιδιαίτερα τις δικές μας αποκλειστικές δικαιοδοσίες. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα μίλησω για τίποτε άλλο, αλλά αυτά είναι οι κεντρικές ιδέες της έκθεσης μου. Αυτά για τα οποία είμαστε αρμόδιοι εμείς. Πρώτον, από πού προέρχονται τα χρήματα. Τονίζω ότι στην έκθεση δεν επικρίνω ή κατακρίνω τη φιλοσοφία ή τη στρατηγική που προτείνει η Κομισιόν να χρηματοδοτείται από τον προπολογισμό δηλαδή η ενωσιακή εγγύηση για αυτά τα ποσά. Παρ' όλα αυτά και άλλα είμαστε πεπισμένοι ότι ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν ταυτόχρονα περικόπτουμε προγράμματα που ήδη αρχίζουν να χρηματοδοτειται απο τον προπολογισμο δηλαδη η ενωσιακη εγγυηση για αυτα τα ποσα παρολα αυτα και αλλα ειμαστε πεπισμενοι σήμερα και γι' αυτό είμαστε αντίθετοι στην προτινόμενη χρηματοδοτική και δημοσιονομική στρατηγική για τη χρηματοδότηση του ΕΦΣΥ. Τα προγράμματα που θα χρηματοδοτεί αυτό το πρόγραμμα δεν θα είναι αποκλειστικά δικά του και άρα για την έρευνα τουλάχιστον αποκλείονται για το λόγο, στην πρόταση της Κομισιόν. Γι' αυτό εμείς προτείναμε κάτι εναλλακτικό. Να αποφύγουμε τις περικοπές για τα υπάρχοντα προγράμματα και βλέπετε ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 έχουμε από αυτού αποκλειστική αρμοδιότητα. Η χρηματοδότηση μπορεί να επιτευχθεί με τις προοδευτικές δημοσιονομικές μας δεσμεύσεις και η διαθεσιμότητα της εγγύησης για την ΕΤΕ θα αρχίσει να ισχύει μόλις τεθεί ενισχύει και η συμφωνία αρχίζει να λειτουργεί το πρόγραμμα δηλαδή, το ταμείο. Κατά την ετήσια εξέταση του προϋπολογισμού είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε όλη την απαραίτητη ευελιξία τα υπόλοιπα, τα περιθώρια του προϋπολογισμού 14, 20 και το πολδίπε βέβαια. Θέλω να τονίσω απολύτως ότι η στρατηγική αυτή δεν είναι μόνο στρατηγική της Επιτροπής μας και της ΤΡΑΝ. Οι εκθέσεις την ίδια στρατηγική δείχνουν Δεν είναι δηλαδή γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε χρήματα εμείς. Την ίδια στρατηγική και στην ΕΚΟΝ και στην ΚΟΜΠΟΥ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα. Δεύτερον, πού θα πάνε τα χρήματα. Ξέρετε τι φρονώ γενικώ ότι πρέπει γενικά οι δαπάνες να συμφωνούν με τα προγράμματα που έχουμε ήδη εγκρίνει όπως τους κλιματολογικούς στόχους κτλ. Άρα πρέπει να επιμείνουμε για τις μεταφορές με λιγότερες εκπομπές και άλλα τέτοια. Θα δείτε ότι τονίζω ιδιαίτερα το θέμα της ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Δεν είναι βέβαια κάτι καθεαυτό πιο σημαντικό από την ψηφιακή οικονομία, αλλά πιστεύω ότι η ενεργειακή αποτελεσματικότητα μας δίνει κάτι παραπάνω κοινωνικά και οικονομικά. Τα έχουμε βέβαια ξαναπεί για τους ενεργειακούς στόχους, αλλά αν δεν τους συμπεριλάβουμε και εδώ τότε δεν θα υπάρχουν αρκετά προγράμματα εξοικονόμησης ή αποτελεσματικότητας ενέργειας. Τα σχέδια που υπέβαλαν τα κράτη-μέλη, από αυτά τα σχέδια μόνο τα πέντε έχουν την έννοια της ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Ενώ η Κομισιόν μας έχει πει ότι πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα και πρέπει και το ΕΦΣΙ να το προβλέπει αυτό. 20% προέβλεψα να έχει το ΕΦΣΙ η εγγύηση του ΕΦΣΙ για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Ξέρω ότι αυτό θα συζητηθεί πολύ, αλλά ήθελα να ξέρετε ότι το θεωρώ πολύ σημαντικό. Τέλος πρόεδρε, να αναφέρω λιγάκι άλλες τροπολογίες. Δηλαδή, πώς πρέπει να γίνονται οι επενδύσεις στην Ένωση, αφού έχουμε το 5-2 και εκεί αποκλειστική αρμοδιότητα εμείς θα αποφασίσουμε ποια θα είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα σχέδια και άρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι What we ότι και η ΕΤΕ θα εφαρμόζει αυτά τα κριτήρια. Ναι. Όλα αυτά βέβαια θα αποφασίζονται καθημερινά από την Επιτροπή Επενδύσεων που πρέπει να αποτελείται από γνωστούς εμπειρογνώμονες και να ασχολείται με τα θέματα που μας αφορούν ιδιαίτερα στο 5-2. Στην έκθεση της οίκων θα δείτε ότι ακούγονται και άλλες ιδέες για τη διακυβέρνηση Αυτές θα τις συζητήσουμε τις επόμενες εβδομάδες ώστε να συμβιβαστούμε σωστά και με αυτούς. Και ξανακαταλήγω ότι στις 13 λίγη ήδη η διορία κατάθεσης τροπολογιών, δεν έχετε πολύ χρόνο λοιπόν. Αλλά είμαι βέβαιη ότι οι τροπολογίες που θα καταθέσετε θα ενδυναμώσουν την έκθεση που έχετε μπροστά σας ιδιαίτερα για την έρευνα και την καινοτομία και την ψηφιακή οικονομία. Επαναλαμβάνω ότι είναι πολύπλοκο το πρόβλημα αλλά δεν έχει νόημα να γνωμοδοτήσουμε απλώς εμείς την Ήτρε, πρέπει να το συνδυάσουμε αυτό και με την Ίκον και με την Τραν. Σας κατευχαριστώ κυρία μου και για τη συνεργασία μεταξύ των τριών επιτροπών τεσσάρων. Ισκιώδης. τέσσερα λεπτά ο καθένας, ένα, το ΕΛΚ. Σας συγχαίρω γιατί είναι πολύ καλή η δουλειά σας και δεν το λέω αυτό από τη συνήθεια ευρωπαϊκή ευγένεια. Πραγματικά το εννοώ διότι η θέση του Κοινοβουλίου και από άποψη της Επιτροπής μας δεν είχε ξανακουστεί τόσο ρητά. Το συνδυάσατε και με τον ορίζοντα ήδη 2020. Νομίζω ότι συμμεριζόμαστε την ιδέα ότι με τη συνεργασία με τις διάφορες επιτροπές θα βρεθεί εναλλακτική λύση για τον προϋπολογισμό. Σας ακολουθούμε λοιπόν σε αυτό, <coughs> αλλά βέβαια όπως φαντάζεστε μπορεί να χρειαστεί και κάποια μικροδιευθέτηση. Δεν αμφισβητούμε λοιπόν την πρόταση θεωρητικά, αλλά στην πράξη αναζητούμε πιο έξυπνες λύσεις. Η κεντρική σας ιδέα πάντως είναι πολύ καλή για το Κοινοβούλιο νομίζω. Παρά όμως ότι τα συμμεριζόμαστε αυτά και για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, ειδικά για αυτό το θέμα, ίσως να πούμε ότι για τη χρηματοδότηση της πρέπει να τονίσουμε και θέματα ενεργειακών υποδομών γιατί είναι διακρατικό θέμα αυτό να τονίσουμε λίγο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενδιαφέρουν τόσο πολύ το κοινοβούλιο. Το άλλο θέμα, άλλα θέματα σχετικά, μήπως να βάλετε τίποτα για να μπει και το RGD στο Διοικητικό Συμβούλιο. για τις προτεραιότητες τώρα το λεγόμενο ER marking. Ίσως να φτάσουμε μέχρι το 25%. Το σημαντικότερο είναι να φανεί πώς θα συνδυαστούν τα υπάρχοντα εργαλεία με το ΕΦΣΙ γιατί έχουμε και άλλα δημοσιονομικά χρηματοδοτικά εργαλεία και δεν πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις εφόσον μάλιστα έχει φανεί από την πρώτη δοκιμαστική φάση ότι μπορούμε να αποφύγουμε επικαλύψεις ώστε το εργαλείο αυτό να δουλέψει αποτελεσματικά και για τις καινοτόμες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες. Αυτό από εμάς και σας συγχαίρω εκ νέου. Σας κατευχαριστούμε. συνόσκι, το Σινόσκι από τους συντηρητικούς. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και την ε, εισηγήτρια στον πολύ λίγο χρόνο που είχε κατάφερε να προετοιμάσει αυτή την ε, έκθεση να συναντήσει τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Γνωρίζουμε σύμφωνα με την εμπειρία μας πως ήταν πραγματικά πάρα πολύ λίγος ο χρόνος που είχε στην ε, διάθεσή της και πραγματικά αξίζει να αξίζει τα συγχαρητήριά μας. Λοιπόν, έχω τώρα εγώ θα έλεγα τέσσερις τομείς ε, που βρίσκω πολύ σημαντικούς. Ε, πρώτον, από πού θα βρεθούν τα λεφτά. Συμφωνώ με την εισηγήτρια πως ε, στον ορίζοντα 2020 και στο... και στο CEF ε, θα είναι πάρα πολύ δυσάρεστο το να παρέμβουμε και να πάρουμε λεφτά από εκεί γιατί είναι ούτως ή άλλως ε, επιστημονικά προγράμματα και πάρα πολύ στοχευμένα. Ένα ερώτημα είναι είναι ότι εάν ε, κάνουμε συνεχώς ε, μεταφορές ε, κονδυλίων ε, από εδώ και από εκεί στον προπολογισμό δημιουργείται μια βεβαιότητα και ίσως δημιουργηθεί ένα προηγούμενο το οποίο το τέλος δεν μπορούμε να ξέρουμε. Εάν τελικά παρέμβουμε και χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα θεωρώ πως χρειάζεται να διατηρηθεί μια συγκεκριμένη δομή όπως είχαμε ακριβώς ορίζει το 2020 και το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Δεύτερον, πού θα πάνε αυτά τα λεφτά. Δεν ε, συμφωνώ απολύτως πως ε, η μοναδική δραστηριότητα θα πρέπει να είναι η εξοικονόμηση της ε, ενέργειας. Τον συζήτησα με την κυρία εισηγήτρια. Υπάρχει και η ενεργειακή ασφάλεια και υπάρχει και ασφάλεια του συστήματος ε, ολόκληρου. Πρέπει να τα έχουμε αυτά κατά νου. Τρίτον, τα κριτήρια επιλογής. Εγώ καταλαβαίνω την πρόταση να εστιάσουμε στην ε, ενεργειακή αποτελεσματικότητα, αλλά αυτό το πρόγραμμα ε, το εξαιρετικό θα πρέπει να εστιαστεί περισσότερο στην ε, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ε, και τα λοιπά. Αυτό το οποίο δηλαδή πάντα προσπαθούμε να πετύχουμε με τις ευρωπαϊκές επενδύσεις. Και βεβαίως τελευταίο έχουμε μία έκκληση για το εξής. Ε, εάν ε, λειτουργήσουν όλα αυτά τα οποία προβλέπουμε εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρξει μια απλοποίηση και να μην ε, επαναληφθούν τα ίδια προγράμματα. Γι' αυτό είμαστε πεπισμένοι πως είναι αναγκαίο το πρόγραμμα αυτό να αποτελέσει μια εξαίρεση να είναι κάτι το οποίο θα γίνει άπαξ και να έχουμε ένα μηχανισμό επενδύσεων για να μην επιβαρύνουμε τους επενδυτές. Έξι δευτερόλεπτα παραπάνω. Ωραία, σας ευχαριστώ. Θα πρέπει να το συζητάμε τα θέματα της βάδας. Ο κύριος Ντεμπάκερ για την Άλντε. Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια. Έκανε τρομερή δουλειά. Όντω δούλεψαν υπό δύσκολε συνθήκε, πάντω νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο. Ότι είμαστε ενωμένοι σε αυτή την υπόθεση, ότι δηλαδή δεν θέλουμε στον ευρωπαϊκό προπολογισμό για το Connecting Euro Facility δεν θέλουμε κάτι άλλο. Θέλουμε να βρούμε κάποιε λύσει δημιουργικέ Να βρούμε τα χρήματα τα οποία χρειάζεται το ΕΦΣΙ για να ξεκινήσει. Γιατί ακριβώ περί αυτού πρόκειται. Έχω κάποιε παρατηρήσει από πλευρά μου. Θα προσπαθήσουμε και εμείς ως Άλντε να βάλουμε το λιθαράκι μας για αυτά τα άρθρα 18 και 19 αποκλειστικής αρμοδιότητας. Το πρώτα πρώτα νομίζω ότι εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει αυτό να το προστατεύσουμε σαν ένα άρθρο ή σαν ε, αιτιολογική έκθεση, αλλά αυτό για να γίνει θα πρέπει να, μην, ε, να καταπολεμήσουμε τις αγορές και την κατάρρυμισή του στην Ευρώπη, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι κεφαλαίοι αλλά και ό,τι άλλο προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρούν ταυτόχρονα. Ιδάλλως τα χρήματα δεν θα ρεύσουν. Πού προέρχονται τα χρήματα. Είναι πάρα πολύ σαφές όταν αρχίσαμε να συζητούμε διάφορες επιτροπές είναι σαφή η στρατηγική είναι σαφές το μήνυμα στα κρατημέλη ζητήθηκαν περισσότερες ε, επενδύσεις τόσα χρόνια. Ε, άρα τώρα είναι δυνατόν να ε, γκρεμίζεται αυτές τις ρήτρε που έχουμε. Πρέπει να υπάρχει ευελιξία στο αποθεματικό πριν ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα και αυτό θα είναι σαφέ το μήνυμα προ κράτη-μέλη και προ ε, Συμβούλιο για να κάνω αυτά που υπόσχονται. Πού θα πρέπει να πάνε τα χρήματα, θα πρέπει να έχουμε ανοιχτό πνεύμα και καταλαβαίνω αυτά που είπε η συγγήτρια για αποτελεσματική χρήση των πόρων. Ναι, αυτό θα πρεπει να πανε τα χρηματα θα πρεπει να εχουμε ανοιχτο πνευμα και καταλαβαινω αυτα που ειπε η συγκιτρια για αποτελεσματικη χρηση των πορων ναι αυτο θα πρεπει να το συζητήσουμε γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο. επίση να έχουμε ευρύτερη προσέγγιση για να λέμε ότι αυτά όλα μπορεί να φυγαμίζονται με το Horizon 2020 και με το Connecting Europe Facility να εξασφαλίσουμε ότι οι εγγύσεις που φτιάχνουμε να καλύπτουν και τα, τις ιδιωτικές επενδύσεις που ήδη έχουν αρχίσει να τρέχουν και στο τοπικό επίπεδο. Επομένω, να μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτούς που ήδη έχουν αρχίσει τις επενδύσεις και μην έχουμε ε, υποκατάσταση, να μην έχουμε διαρροές και να συνεργαστούμε με το επενδυτικό ταμείο και την επενδυτική τράπεζα. Εγώ θέλω να σας πω ότι θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση λογοδοσίας. Λένε τα κράτη-μέλη, ας δώσουμε όσο γίνεται περισσότερες αρμοδιότητες σε τράπεζα και επενδυτικό ταμείο. Μα έτσι όμως ε, αφαιρείται η δυνατότητα του Κοινοβουλίου να εμπλακεί. Δεν λέω ότι δεν εμπιστεύουμε τους επαγγελματίε, αλλά θα πρέπει όπως σε κάθε επένδυση να μιλούμε στους ε, μετόχους που θέλουμε να έχουμε και να τους εξηγήσουμε τι γίνεται, να τι πάνε να πει υποχρέωση λογοδοσίας. Αλλά, άρα να μην θεωρούμε ότι δεν υπάρχει εδώ πέρα τίποτα το ιδιαίτερο και ότι δίνουμε επιταγή λευκό στην ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα πρέπει και πάλι να γίνει η Ευρώπη ελκυστική για τις ξένες επενδύσεις. Τώρα, αυτά τα πρεσβεύει η πολιτική μου ομάδα και ελπίζω ότι θα τα βρούμε τελικά. Και τελικά θα γίνουμε ανταγωνιστικοί και θα μας σε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ ο κύριος για τους πρασίνους. Σας ευχαριστώ. Και εγώ όπως ε, και οι άλλοι συνάδελφοι θεωρώ ότι η συγκίτρια τα πήγε πάρα πολύ καλά. Άρα θα πρέπει να είμαστε στρατηγικοί, θα πρέπει να έχουμε μια θέση ενωτική, όλο το κοινοβούλιο μας ε, υποστηρίξει και να μπορούμε να έχουμε μόχλευση στις διαπραγματεύσεις. Μπράβο στην Εγώ Τα ξεστρέφουμε στις πράσινες να υπάρχει προσθεμένη αξία, να υπάρχει υλοποίηση της πολιτικής του 2020. Σας ευχαριστούμε που αυτά τα ξεκαθαρίσατε στο κείμενο σας. Επίσης, τα διασυνοριακά, όλες οι υποδομές θα πρέπει να εμπλακούν, να χρησιμοποιηθούν και για το crowding out. Εάν έχουμε το connecting facility για την ενέργεια και τις μεταφορές, τότε υπάρχει πιο σημαντική εγγύηση ότι θα έχουμε διασυνοριακή ρύθμιση για αέριο, για ηλεκτρικό, για δρόμους, για οδικές μεταφορές. Αλλά να μην απονευρώσουμε το Ταμείο γιατί μην κάνουμε το λάθος να μην αλλάξει τίποτα. Μιλούμε για το Συνδέοντα την Ευρώπη ότι δουλέψαμε τρία χρόνια. Άρα αυτό το οποίο κάναμε το διαφυλάξουμε. Είναι μια υπόσχεση που να την τηρήσουμε. Τώρα για την τεχνική βοήθεια. Θα πρέπει να γίνει αυτό με πρωτοβουλίες αποκεντρωμένες. Με τα πανεπιστήμια, με τις νεοφυείς επιχειρήσεις, με τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου. Όλα αυτά να καλυφθούν για την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Ευχαριστούμε που το θίξατε. Μην το μιλάμε για να δώσουμε δουλειά στους Καλιφορνίους και στους Κινέζους. Είναι δουλειά για τους Ευρωπαίους. Οι συμβάσεις θα αφορούν ακριβώς αυτή τη χρήση της ενέργειας. Έχουμε δύο ταμεία. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και το Ελλήνα τεχνικής αρρωγής. Μιλάμε για 200 ε, δις επενδύσεων σε Βαρκελόνη, στο Μιλάνο. Έχει ελκύσει τρομερές επενδύσεις. Να η μόχλευση. Και με το Ταμείο Ανασυγκρότησης. Και με το Ταμείο Εποτεχνικής Ενέργειας. Το κάνει η Deutsche Bank. Το διαχειρίζεται. Μιλάμε για 200 δις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Βλέπουμε ότι η ενεργειακή αποτελεσματικότητα είναι καλή για την οικονομία, αλλά απεδείχθη ότι αποτελεί και μια πολύ σημαντική μόχλευση. Και επεμπιπτόντως θα βοηθήσει την Ανατολική Ευρώπη όσον αφορά την κρίση με τη Ρωσία. Γιατί είναι κρίση θέρμανσης, κρίση φυσικού αερίου. Οπότε τα μέτρα αποτελεσματικής ασφάλεια είναι αυτό που χρειάζεται η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία και η Πολωνία. Αυτό χρειάζεται. Οπότε με περισσότερη αποτελεσματικότητα θα ενώσουμε την Ευρώπη ενεργειακά γιατί για το ίδιο ΑΕΠ η Ανατολική Ευρώπη ε, αναλώνει ενέργεια 2, 3, 5 και παραπάνω φορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Λόπες Μπερμέχο. Από την ΚΟΕ θα μιλήσει αργότερα, θα έρθει αργότερα γιατί είναι στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πρώτα. Πρώτα πρώτα ευχαριστώ στην κυρία Φάνμπερτ γιατί πάρα πολύ αξιόλογη ήταν η δουλειά της, ενώ είχε λίγο χρόνο στη διάθεσή τη. Και επίση ε, συμφωνώ 100% για το ότι δεν είναι σωστέ αυτέ οι περικοπές για το 2020. Γιατί θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά την αριστεία στην Ευρώπη. Και αναφέρουμε το πρόγραμμα Μαρία Κιουρί. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς στον προϋπολογισμό θα βρούμε τους πόρους χωρίς αυτό είναι τόσο περίπλοκο γιατί κάθε χρόνο υπάρχει πρόβλημα στο σκελισμό του προπολογισμού. Άρα χρειαζόμαστε και πια εναλλακτικά, εναλλακτικού πόρου. Ε, αλλά για να μην περικοπούμε το ορίζον 2020. Ως εναλλακτική λύση έχουμε του πόρου του προενταξιακού. Μα το είπε αυτό και η Επιτροπή Γιούνγκερ πριν από λίγους μήνες και ότι θα το κάνει αυτό με το 2019. Να, σήμερα είμαστε σε κάποιο λεπτό σημείο. Οπότε να μην παίρνουμε πόρους από αυτά τα οποία ε, αναθερμαίνουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Είπαμε επίσης ότι θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις στην πράσινη οικονομία για να πετύχουμε τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους, ιδίως όσον αφορά την ε, αποτελεσματική χρήση ενέργεια. Μην ξεχνούμε ότι έτσι έφτιαξε ο Γιούγκερ το πρόγραμμα για να βγει η Ευρώπη από την σοβαρή αυτή κρίση. Σε κάποιες χώρες, σε κάποιες περιφέρειες, ολόκληρα κομμάτια του πληθυσμού πέσανε στη φτώχεια. Άρα να τους βοηθήσουμε αυτούς, αυτούς που έπληξε περισσότερο η κρίση. Και θα πρέπει να δούμε με τι μηχανισμός θα βοηθήσουμε επενδύσεις σε αυτές τις περιφέρειες που έχουν πέσει και μειωθεί οι επενδύσει. Άρα θα πρέπει να βρεθεί ένα τέτοιο μηχανισμό. ε, αλλά προσοχή μην αυξηθεί το χάσμα μεταξύ ε, των περιφερειών που έχουν πληγεί των υπολείπων. Τέλος πάντων έχουμε και άλλες τροπολογίες και εμείς είμαστε υπέρ όλων των μέτρων που θα βοηθήσουν τις επενδύσεις για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, για ε, την έρευνα και για τις ΜΜΕ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ συνάδελφε. Okay. Shall we go to, to other speakers? Let's say Πάμε τώρα στου επόμενου ομιλητέ. Παρακαλώ μην μιλήσετε πάνω από τρία λεπτά. Άντε, δυόμιση. Ταμπουράνο είναι ο πρώτο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Αποκλίνει ε, ε, αυτό το οποίο λέει από την ε, Επιτροπή και άλλα και εμείς συμφωνούμε. Όπως τα είπε και ο κύριος Μπορέλη. Πρέπει να σας πω ότι όντως αυτή η πόρη για την προενταξιακή πορεία ιστορικά, κάτι γνώμη μου, ήταν ένας αναχρονισμός και άρα θα πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε υπέρ όσων έχουν τώρα οικονομικά στριμωχτεί. Μεγάλη δυσκολία παίρνουν τώρα οι μικρές επιχειρήσεις, πιο πολύ από τις μεσαίες, λόγω της κρίσης της πιστοτικής. Δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί για να τις ε, καλύψουν. Μιλώ για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, τις παραδοσιακές, τις βιοτεχνίες. Και ιδίω στην Νότια Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικέ αυτέ οι επιχειρήσει για τον κοινωνικό ιστό. Ευχαριστώ, συνάδελφε, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επισημάνω τα επιχειρήματα που θα αντιτάξει η Κομισιόν όταν ακούσει την κριτική μας για το διαγούμισμα του προπολογισμού του 2020 θα πούνε πως ε, η οικονομική δραστηριότητα που θα προκαλέσει το πρόγραμμα αυτό επενδύσεων θα προκαλέσει ανάπτυξη και επενδυτικές δραστηριότητες που θα αντισταθμίσει ε, αυτά τα οποία αφαιρούμε από τον προϋπολογισμό του 2020. Εγώ πέρασα όλη μου τη ζωή στη βιομηχανία, στην έρευνα κτλ. και έχω μάθει το εξής πως οι εταιρείε δυσκολεύονται πάρα πολύ να επενδύσουν σε έργα τα οποία είναι τόσο μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα του καπιταλισμού οπωσδήποτε. Γι' αυτό όλες οι καπιταλιστικές χώρες ε, φορολογούν τις εταιρείε ε, και μετά με τους φόρους αυτούς χρηματοδοτούν ερευνητικά προγράμματα. Οπότε σας ζητώ να μην δεχτείτε το επιχείρημα αυτό της ε, Κομισιόν. Μπορεί πράγματι να έχουμε περαιτέρω ανάπτυξη στην βιομηχανία, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να αντισταθμίσει την μακροπρόθεσμη έρευνα. Σας ευχαριστώ. Σαφχάουζερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για αυτή την έκθεση που όπως το είπαν και άλλοι είναι πολύ καλή δουλειά. Εγώ μιλώ ως παλαιός πρώην υπεύθυνο για την ενέργεια στην περιφέρειά μου την Αλσατία. Από πού προέρχονται τα χρήματα ρωτήσατε. Νομίζω ότι το θέμα πρέπει να τεθεί. Το καντιτά, την ποσοτική χαλάρωση να μην την easing που λέμε και εμείς. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούμε όποτε μπορούμε το νομισματικό εργαλείο. εργαλείο. Να τοποθετούμαστε, να μην χρησιμοποιείται μόνο για, να μην εξυπηρετεί μόνο τις τράπεζες αλλά και την πραγματική οικονομία. Τώρα, το ότι χρησιμοποιούμε θέσεις του προϋπολογισμού γιατί όχι, γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε θα έλεγε κάποιος τα ταμεία που δεν πολύ χρησιμοποιούνται, τα ταμεία για τη, τις θέσεις για τη διεύρυνση, ας πούμε αφού δεν προβλέπεται διεύρυνση. Αλλά ούτως ή άλλως εδώ αναλαμβάνεται ένα τεράστιο στίχημα από την Κομισιόν και τον κύριο Γιούνκερ μέσω εγγυήσεων δηλαδή να κινητοποιήσουμε μακροπρόθεσμα επενδύσεις που δεν θα γίνονταν χωρίς αυτές τις εγγυήσεις. Θα βρεθούν όμως σχέδια. Πού θα πάει τώρα το χρήμα. Η πιο σίγουρη επένδυση σήμερα είναι στην ε, ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Παράδειγμα που πολλές φορές το έχουμε πει. 400 δισεκατομμύρια εισαγωγών. Αν και μόνο 10% από αυτά εξοικονομηθούν θα έχουμε 40 δισεκατομμύρια. Επομένως δεν θα αρκούσε ούτε καν όλο το σχέδιο Juncker για να εξισορροπήσει για να φέρει το ίδιο χρήμα με μια απλή εξοικονόμηση ενέργειας. Πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει όμως αποκεντρωμένα. Πρέπει να παίξουν τα κράτη αλλά ακόμη περισσότερο οι περιφέρειές των και οι τοπικοί παράγοντες Γι' αυτό δεν είναι απαραίτητα σωστό ή έξυπνο να λέμε ότι για την Ελλάδα ας πούμε η γαλλική ΔΕΗ θα συνδεθεί αποτελεσματικά και υποχρεωτικά με τους παράγοντες αυτούς τους τοπικούς. Τώρα, πού πρέπει να πάνε τα χρήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εκείνες που πραγματοποιούν τις εξοικονομήσεις. Αλλά ξέρουμε από εμπειρία ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη συμπερίληψη στα σχέδια αυτά των αποκεντρωμένων παραγόντων, των τοπικών δηλαδή παραγόντων. Και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τοπικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ευχαριστούμε. Κυρία Καμπεσόν Λουίς. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εγώ συγχαρώ την κυρία Φαν γιατί έδειξε θάρρος και πραμήθηκε το Horizon 2020 για αυτόν τον προπολογισμό και πέτυχε και μια θέση συνενετική εδώ και παράξω και για τις άλλες εμπλεκόμενες επιτροπές. Οι σοσιαλιστές επιθυμούν φιλόδοξες επενδύσεις, αλλά δεν θέλουμε να χαλάσουμε ό,τι φτιάξαμε για να κάνουμε κάτι καινούργιο. Θέλουμε την οικονομική ανασυγκρότηση στην Ευρώπη και με το πρόθεσμα για να γίνει αυτό χρειάζονται υγιείς, εύρωστες επενδύσεις. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να συνεχίσουμε και να υλοποιήσουμε ένα τέτοιο σχέδιο επενδύσεων. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει στον κανονισμό να υπάρχει ως προϋπόθεση ε, αυτό το ποσοστό για όλα τα προγράμματα και έργα τα οποία αφορά το ΕΦΣΕ. Για κάθε χρηματοδότηση να έχουν σχέση με καινοτομία, με τεχνολογία, με τα κέντρα έρευνας, αλλά επίσης και να υπάρχει κρατική προμήθεια καινοτόμου τεχνολογίας. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτά τα οποία θέλει η Κομισιόν, τα οποία είναι συντηρητικά. Θέλει να αφήσει απ' έξω ολόκληρο τομέα, γιατί η καινοτομία και η έρευνα περνούν από επένδυση και σε ανθρώπινους πόρους. Και βέβαια είναι αλήθεια ότι θα πρέπει και αξίζει να ρισκάρουμε περισσότερο από σε Με το ΕΦΣΥ θέλουμε την ε, αναθέρμανση της ευρωπαϊκής οικονομίας Θέλουμε να δημιουργήσουμε απασχόληση, αλλά επίσης θέλουμε και να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ με την εμπλοκή τους σε αυτή την υπόθεση. Πρόεδρος, εκτός μικροφώνου. Ναι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για επόμενη ομιλία νομίζω ότι η Κάτσελα έκανε δουλειά πάρα πολύ θετική, ε, αλλά επίσης έκανε και ε, μια στέρεη αρχή για να εξετάσουμε τα πράγματα και θα ήθελα να πω στη συνέχεια το για αυτά τα τρία λεπτά που έχω ότι είναι πολύ σημαντικό νομίζω αυτό το οποίο προτάθηκε και το οποίο έχει να κάνει με τα όσα είπε και η Επιτροπή Οικονομική και η Μεταφορών το πώς θα αλλάξει η βάση της χρηματοδότησης γιατί είναι τελείως παράλογο το να πάρουμε χρήματα από την έρευνα και την τεχνολογία. Ε, έτσι στηρίζονται τα προγράμματα και τα έργα. Και επίσης με μεγάλη προσοχή θα πρέπει σε συνεργασία με την ε, εισηγήτρια να βρούμε κάποιες εναλλακτικές. Αλλιώς όλα αυτά τα οποία είπαν για για την, ε, για την έλλειψη χρημάτων, για τη στέρεη βάση που πρέπει να έχουμε, όλα αυτά να, να μην τα χάσουμε. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε για να μην απονευρώσουμε την πρόταση. Υπάρχει το θέμα το οικονομικό και πρότεινε κάποια οικονομικά μέτρα ε, η Επιτροπή, η Επιτροπή Οικονομική για τις οφειλές ε, και για τις σχετικές ρήτρες όμως να μην θέσουμε εν κινδύνο εκείνες τις χώρες που ήδη ίσως κέλυσαν δύσκολο τον προπολισμό, μην ξαναπέσουν στο πρόβλημα. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μια κρατική τράπεζα, αλλά όταν δεν γίνεται αυτό να έχουμε κάποια, κάποια που οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη. Επίσης, οι τομείς αναφορά θα πρέπει να είναι εκείνοι οι τομείς οι οποίοι κλαρσίκωση ενέργεια, ενέργειας, τα ψηφιακά, η ανάπτυξη της τεχνολογίας για τις ε, επιχειρήσεις, μεταφορά τεχνολογίας, γιατί αυτό στην Ευρώπη είναι αιτία ανισοτήτων όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα γιατί έχουμε ζώνες, περιοχές, χώρες λιγότερο ανταγωνιστικές από άλλες γιατί έχουμε αυτή τη μεταφορά τεχνολογίας. Άρα εκεί θα πρέπει τώρα να προσέξουμε. Και να δούμε τι γίνεται και σε, από πλευρά της παιδείας, προετοιμασίας ανθρωπίνων πόρων, όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν προτεραιότητες. Ο δεύτερο λόγος, ρόλος του Κοινοβουλίου. θα Συμμετάσχουμε και εμείς με κάποια κριτήρια και να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε υποπτία και έλεγχο για την επιλογή των προγραμμάτων. Όχι, να μην έχουμε επικάλυψη αν πρέπει άλλος να κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά ούτε πρέπει να είμαστε απόντες από αυτή τη διαδικασία του ελέγχου που είναι και δική μας αρμοδιότητα. Ροντρίγκες Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εγώ να αρχίσω με συγχαρητήρια προς την εισηγήτρια άριστη η δουλειά της και πάρα πολύ αξιόλογες οι βελτιώσεις που κατόπιν επέφερε. Έχουμε κάποιες τροπολογίες υποβάλει για να μπορέσουμε να έχουμε την εγγύηση προσβασιμότητας από τις ΜΜΕ στη χρηματοδότηση. Τι λέει η Κομισιόν. Λέει για 3.000 εργαζόμενους. Μα αυτό δεν είναι. Δεν καλύπτει τις ε, ΜΜΕ πρέπει να υπάρξουν και ότι θα πάρουν χρήματα οι ΜΜΕ με την τροπολογία να δοθεί ορισμό να υπάρξουν κριτήρια για το τι είναι ΜΜΕ και εμεί όλοι συμφωνούμε να μην πάρουμε λεφτά από το 2020 ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε χρήμα στην καινοτομία κάτι άλλο που λείπει νομίζω για να προβληματιστούμε. Πρώτον, πολύ εύστοχη εκείνη η τροπολογία που λέει για την οικονομική προσθέμενη αξία και την κοινωνική προσθέμενη αξία. Αλλά θα πρέπει σε όλο το έγγραφο να ενσωματώσουμε διάφορα στοιχεία κοινωνικής πολιτικής. Γιατί όντως θα πρέπει να υπάρξει απόδοση των επενδύσεων οικονομική, αλλά θα πρέπει να γίνεται και δουλειά στο κοινωνικό επίπεδο από πλευρά των επενδύσεων. Άρα να κάτσουμε και να σκεφτούμε πώς θα βελτιώσουμε την κάλυψη κάποιων προγραμμάτων που αναδεικνύουν τις κοινωνικές μας αξίες και τις επιχειρήσεις που βοηθούν σε αυτό την κατεύθυνση και να δημιουργείται απασχόληση εκεί που χρειάζεται και υπάρχουν δυσκολίες. Άλλο. Όσον αφορά την επιλογή των προγραμμάτων επένδυσης, έχουμε μία πάρα πολύ πλήρη τροπολογία. Μπράβο στην συγκεντρία για τα κριτήρια της αξιολόγησης. Θα ήθελα όμως εκεί να προσθέσουμε το ότι θα πρέπει να δημοσιοποιούνται για το ποια προγράμματα απορρίπτονται. Να ξέρει ο κόσμος γιατί απερίφθη ένα πρόγραμμα. Άρα και η αποδοχή και η απόρριψη. Να είναι γνωστά. Να, τι πάει να πει διαφάνεια. Τέλος δε, ε, επίσης είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα κριτήρια επιλογής των εμπειρογνωμών στις σχετικές επιτροπές, στις επιτροπές των επενδύσεων, γιατί αυτοί πρόκειται να αξιολογήσουν τα προγράμματα που θα υποστήξουν τα κράτη-μέλη και τα οποία θα αποδώσουν. Άρα να είναι ξεκάθαρο με τι κριτήρια επιλέγονται αυτοί που θα αξιολογήσουν. Και να δημοσιοποιεί επίσης και τα απορριφθέντα έργα και προγράμματα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να εκτιμήσω, να εκφράσω την εκτίμησή μου για την έκθεση αυτή, για την εισήγηση αυτή. Μερικά σχόλια. Για μένα ο κύριος στόχος του σχεδίου Γιούνκερ είναι η επανάκτηση της εμπιστοσύνης. Έτσι πρέπει να δούμε το θέμα. Μερικοί συνάδελφοι τόνισαν και δικαίως ότι το σχέδιο Γιούνκερ έχει τρία θεμέλια Υπάρχει το δημοσιονομικό, υπάρχει όμως και το θεμέλιο της εσωτερικής αγοράς και το τρίτο για το διοικητικό άχθος είναι επίσης σημαντικό. Θα ήθελα εγώ να τα τονίσω και τα τρία λοιπόν. Μιλάμε για ιδιώτες επενδυτές, για το ότι θα θέλαμε να μειώσουμε την, το έλλειμμα που έχουμε στις ιδιωτικές επενδύσεις. Άρα οι επενδυτές τα λεφτά τους τα έχουν κάπου στι τράπεζες ή οπουδήποτε και πρέπει να τα βγάλουν από εκεί και να τα επενδύσουν. Και αυτό είναι θέμα εμπιστοσύνης αλλά επίσης και σημαντικός λόγος να τους ακούσουμε. Τι επενδύσεις θα ήθελαν να κάνουν. Να δούμε και θέματα δημοσίου συμφέροντος και επενδυτών. Ε, είναι και αυτός ένας λόγος για τον οποίο καλώ την εισηγήτρια να δει τα πράγματα ευρύτερα, όχι μόνο ή κυρίως την αποτελεσματικότητα, ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Αν και αναγνωρίζω τη σημασία της. Ευρύτερα, ευρύτερα. Η Σαμπίνα έκανε μερικά σχόλια και για το ορίζον. Συμφωνώ και με αυτό. Ήμουν και εγώ από τους υπεύθυνους του προγράμματος και πιστέψτε με μερικά τέτοια σχέδια δεν θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Γιούνκερ δεν θα χρηματοδοτηθούν γιατί δεν θα υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον ένας ακόμη λόγος λοιπόν για τον οποίο πρέπει να διατηρηθεί και το Horizon. Τώρα πού να πάνε τα χρήματα εδώ θα εκτιμούσα ιδιαίτερα αν τονίζαμε όχι μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά αν δείτε το σχέδιο του Ταμείου δεν αναφέρεται τίποτα και για τις καινούργιες επιχειρήσεις, τις λεγόμενες startup. Να δοθούν κριτήρια δηλαδή και σε ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση αντί να πάνε στις Ηνωμένε Πολιτείες να έχουν την εμπιστοσύνη να κάνουν την επιχείρησή τους στην Ευρώπη. Ειδική κατηγορία για τις startup δηλαδή. Ένα τμήμα από τα χρήματα για τις μικρομεσαίες να αφορά τις startup. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε συνάδελφε. Τώρα ο σκιώδης της Γκουε, η κυρία Λόπεθ Μπερμέχο, ήρθε και θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, συγγνώμη που καθυστέρησα, γιατί ήμουν στην Ολομέλεια. Και τελικά καθυστέρησα περισσότερο από ό,τι περίμενα εκεί. Άρα, πέραν τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να δώσουμε για τι επενδύσει, αυτό το οποίο θέλουμε εδώ να κάνουμε είναι, κατά τη γνώμη μα, αυτό που θέλουν να τις μειώσουν και αυτό θέλουν να κάνουν περικοπές στον προπολογισμό σημαντικά ούτως ώστε να μην μπορέσουν να τονώσουν τη ζήτηση και να αλλάξουν την παραγωγική βάση. Δεν έχει νόημα ε, αυτές οι υποδομές του Connect, ε, Connecting Europe ή το Horizon 20.000 ε, να πάνε και να βοηθήσουν αυτές τις ε, επενδύσεις ιδιωτικέ, και έτσι δεν μπορεί να υπάρχει από πλευράς δημοσίου ο σχετικός έλεγχος εμείς πάντως ε, χαιρετίζουμε την απόπειρα της ε, ε, εισηγήτριας για να ελέγξει αυτή την κατάσταση με τις περικοπές. Αλλά προσοχή, θέλουμε να γίνει τροποποίηση του κειμένου, να το βελτιώσουμε όσο γίνεται. Αλλιώς δεν θα βοηθήσει τα προβλήματα των Ευρωπαίων. Θα παροξύνει τα προβλήματα. Οπότε είμαστε υπέρ της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. Θα δώσουμε τη μάχη μας για διαφάνεια στις αποφάσεις. Να προσπαθήσουμε κάθε πρόγραμμα να οδηγεί σε συνοχή και απασχόληση. Και επίσης να τηρηθούν οι περιβαλλοντικές διατάξεις. Να γίνεται έλεγχος τέτοιος πριν εγκριθεί. Κάθε σχέδιο. Αν ωφελούνται οι να κοιτάμε. Και τελικά να μην ε, χρηματοδοτείται το πρόγραμμα Juncker από τις τσέπες των Ευρωπαίων φορολογουμένων αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρξουν εγγύησεις ε, αλλά βέβαια δεν τις χρειάζονται επενδυτές οι οποίοι θα πλουτίσουν από τις επενδύσεις. Πρόκειται για ένα μέσο πολιτική το οποίο θα πρέπει η Επιτροπή με τη θέση της να το ενισχύσει. Thank you very much. Uh, Mr. Ευχαριστώ κύριος Ζωρίνιο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα να ξεκινήσω με κάτι γρήγορο επί της ε, διαδικασίας. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση, από τις σημαντικότερες στην Επιτροπή μας και νομίζω πως ε, δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε διερμηνία σε κάποιες γλώσσες. Βλέπω άδεια την πορτογαλική καμπίνα και πολλές καμπίνες είναι άδειες και θα ήθελα να το πω αλλά το σημαντικότερο είναι να υπογραμμίσουμε και την ε, δουλειά που έχει κάνει η Κατλίν ε, και οι υπόλοιποι σκιώδεις εισηγητές ε, και υποστηρίζω βεβαίως την ιδέα να μην στέλνουμε αντιφατικά μηνύματα στην κοινωνία. Πρέπει να υπάρχει κάποια συνέργεια με το εργαλείο αυτό και είναι κρίμα να στέλνουμε όπως είπα μηνύματα αντιφατικά. Το μέσο αυτό για να επενδύσουμε στο μέλλον της Ευρώπης είναι μια πάρα πολύ θετική ιδέα που πραγματικά κινητοποιεί τον κόσμο. Το βλέπω όταν μιλάω μαζί τους για να προετοιμαστεί η Ευρώπη για το μέλλον. Αλλά εάν εμείς ε, κάποια στιγμή κάνουμε περικοπές ε, στην έρευνα, την ανάπτυξη, τον ορίζοντα 20-20 κτλ. Ε, χάνουμε την αξιοπιστία μας και βεβαίως την συνέργεια την οποία θέλουμε να επιτύχουμε. Τώρα συζητάμε κάποια δημοσιονομικά εργαλεία, αλλά το σημαντικότερο είναι αυτά τα εργαλεία. Είναι το όραμα το οποίο υποστηρίζει αυτά τα εργαλεία και νομίζω πως η έννοια αυτή της Ενεργειακής Ένωσης, της Ψηφιακής Ένωσης θα μπορούσε να διαμορφώσει την οικονομία μας και την ικανότητά μας να ανταγωνιστούμε στον κόσμο. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση και πηγαίνει βεβαίως ε, κατευθείαν στην ουσία. Κατά την άποψή μου λοιπόν είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε την ιδέα της ε, δικτύωσης ε, να συνεργαστούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, καινούριες επιχειρήσεις, διάφορα θεσμικά όργανα, θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες έτσι ώστε να μην έχουμε μόνο την ενεργειακή αποτελεσματικότητα αλλά και κάποια αποτελεσματικότητα ως προς την ποιότητα που νομίζω πως λείπει από την έκθεση. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι για όλη τη συζήτηση. Συνήθως υπάρχουν όλες οι γλώσσες αλλά δεν είναι πάντα ε, δυνατόν σε έκτακτες συνεδριάσεις. Τις τακτικές είναι εγγυημένο αυτό αλλά όχι για τις έκτακτες. Rubik Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα βεβαίως να δώσω συγχαρητήρια για αυτή την ε, έκθεση γιατί εγώ αναρωτιέμαι συνεχώς ε, ως μέλος ε, της Επιτροπής Προπολογισμού τι γίνεται με τις πληρωμές, τις δεσμεύσεις, τις προθεσμίες. Αντιλαμβάνομαι πως βραχυπρόθεσμα πρέπει να διαθέσουμε κονδύλια για να μπορέσει να ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό. Μεσοπρόθεσμα όμως πρέπει να σκεφτούμε μήπως οι περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ε, είναι ότι πιο θετικό. Βλέπουμε πως ε, είχαμε πάλι μια ε, νέα περικοπή 4% και 1% στο προϋπολογισμό και πάλι νέες ε, περικοπές προγραμματίζουμε τώρα. Να δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και θεωρώ πως η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς είναι να φτιάξει διασυνοριακές ε, δομές και θα πρέπει παραδείγματο χάρη να ε, δούμε τι γίνεται με την δυνατότητα δημοπράτησης αδειών κινητής τηλεφωνίας. Τα λεφτά αυτά τα οποία είναι δισεκατομμύρια δεν μπορεί να πηγαίνουν μόνο στα χρέη των κρατών μελών αλλά και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν έργα για να, για να χρησιμοποιήσουν και τα δικά τους ε, τα κονδύλια και τα, τρα... και τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Όταν ακούμε εδώ πέρα δηλαδή νούμερα δισεκατομμυρίων ε, που προβλέπονται για τις ε, άδειες νομίζω πως ε, θα μπορούσε κάτι να πάει στον ευρωπαϊκό προπλησμό και να δημιουργηθεί ένας ενάρετος όπως λέγεται κύκλος κάτι το οποίο είναι αναγκαίο, αλλά σοχεύουμε μόνο, όπως είπα, βραχυπρόθεσμα. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και μέσω μακροπρόθεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ αγαπητέ συνάδελφε. Ο κύριος Χέλμερ είναι ο επόμενος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σημειώνω ότι εδώ κάνουμε αυτό το που συνήθως κάνει καλύτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή συζητάει πώς να ξοδέψει όλο και περισσότερα χρήματα των φορολογουμένων. Με ιδιαίτερα με εντυπωσίασε ο τίτλος της παραγράφου 3 ας μην επιμείνω στην φτωχή σύνταξη και έκφραση αλλά θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για το θάρρος της και χρησιμοποιώ τη δική της φράση γιατί τόνισε την επική αποτυχία της μέχρι τώρα πολιτικής για την ενέργεια. Εγώ αυτό το λέω εδώ και πολύ καιρό και είναι πολύ ικανοποιητικό για μένα να βλέπω ότι και κάποιος άλλος συμφωνεί. Παρ' όλα αυτά θα έλεγα ότι δεν έχει τίποτα η γνωμοδότηση αυτή που να λύνει το πρόβλημα. Φυσικά η ενεργειακή αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα είναι κάτι καλό, αλλά και οι ανταγωνιστές μας έχουν τέτοια προγράμματα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε ότι καθεαυτήν η ενεργειακή αποδοτικότητα θα βελτιώσει οτιδήποτε. Εμείς στην Ευρώπη έχουμε στρέψει τα νότα σε χαμηλού κόστους και αποδεδειγμένες τεχνολογίες όπως τον άνθρακα για να επενδύσουμε τις αβέβαιες ε, ανανεώσιμες λεγόμενες ενεργειακές πηγές. Και φυσικά όλα αυτά είναι πολύ πιο ακριβά από ό,τι για τους ανταγωνιστές μας. Ο Σκιώδης από τους φιλελεύθερους μίλησε για τη σημασία που έχει η έλκυση επενδύσεων στην Ευρώπη από αλλού αλλά με τις ενεργειακές τιμές που έχουμε δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο γιατί οδηγούμε την απασχόληση και τις επενδύσεις και την βιομηχανία εκτός Ευρώπης και πολλές από αυτές τις βιομηχανίες θα πάνε αλλού όπου υπάρχουν χαμηλότερα κριτήρια προστασίας του περιβάλλοντος. Υπονομεύουμε λοιπόν την ανταγωνιστικότητα και διώχνουμε τις επενδύσεις και την απασχόληση. Και παράλληλα δεν μειώνουμε, δεν καταφέρουμε να μειώνουμε τις εκπομπές διοξιδίου. Αυτή είναι η επική αποτυχία. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπω τίποτα στην γνωμοδότηση που να το λύνει. Ευχαριστούμε. Τσαμανάτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θεωρώ ότι η Κάτλα έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν και είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά όλα αυτά τα οποία λέει ούτως ώστε να μπορούμε να προστατεύσουμε τους πόρους που χρειάζεται να πάνε για ε, την υπόθεση αυτή να μην από το ορίζον 2020 να πρέπει να πάνε προς κάποιες κατευθύνσεις στρατηγικές και πιο συγκεκριμένα να πάνε ε, στην υπόθεση της αποτελεσματικής της ενέργειας. Τώρα υπάρχει κάτι άλλο το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να τονιστεί. Ε, θέλω να σας πω για όλα ε, αυτούς τους περιορισμούς που αναφέρθηκαν όλους αυτές τις περικοπές γιατί πολύ περισσότερο έχουν επενδύσει οι Αμερικανοί και για τον ΦΠΑ που είναι τόσο υψηλός αυτά δεν είναι αξιόπιστες λύσεις αλλά επίσης αυτό αφορά και ε, κάποιον ε, μηχανισμό ο οποίος ε, έχει εξατομικευμένη φύση για κάθε επένδυση, κάτι το οποίο θα είναι επιβραδυντικός παράγον. Επομένως αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να λειτουργεί το σύστημα. Χρειάζεται να μην βάζουμε σε κίνδυνο το εύση. Για μένα αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να αναλάβουμε. Ότι θα πρέπει αυτό να ανατονιστεί. Ότι είμαστε σε κατάσταση κατά την οποία οι πόροι οι οποίοι θα εκταμιευτούν για τις ε, ε, επενδύσεις δεν θα επιβαρύνουν τόσο πολύ. Επίσης θα πρέπει να καταλάβουμε τι γίνεται με το ΦΠΑ. Θα πρέπει επομένως να μην πούμε στον ιδιωτικό τομέα σου δίνουμε ένα ευρώ και εσύ να επενδύσεις 15 και θα σου πούμε πώς θα το κάνεις αυτό. Θα πρέπει να του έχουμε ήδη καλύψει. Θα πρέπει να επισημανθούν οι κίνδυνοι. Αλλιώς δεν θα υπάρξει συμφωνία. Επομένως θα πρέπει να, μην, να υπάρξει χρηματοδότηση αρκετή και όχι υποχρηματοδότηση. Γιατί αλλιώς δεν θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε, δηλαδή να έχουμε ιδιωτικό κεφάλαιο 15 πλάσιο του δημοσίου, του κρατικού. Άρα προσταθήκατε τα αυτή επενδύσει. Και επίσης μετά έχουμε εδώ κάποια όρια, ε, δηλαδή το πόσα χρήματα έχουν τα κράτη-μέλη. Να βρεθεί επομένως ένας τρόπος ε, ισοσκελισμού των προϋπολογισμών χωρίς να παραβλάψουμε την προϋποδότηση του ορίζον 2020. Γι' αυτό σας λέω ότι θα πρέπει πάνω σε αυτό να δουλέψουμε να δούμε τι γίνεται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα πρέπει να μπορούν να ωφεληθούν από τις επενδύσεις και άρα θα πρέπει να βρούμε και άλλα μέσα πολιτικής. Αλλιώς ε, κινδυνεύουμε να κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Να μείνουμε δηλαδή με τις προσπαθίες μας μόνο με τον ενθουσιασμό. Μίριαμ Τάλι. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου και εγώ να συγχαρώ την Κατελάνη για την ε, γνωμοδότηση της τη διάβασα και συνδυάζει πολλές ιδέες δηλαδή μπροστά μας έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε τις διαφορετικές αυτές μεταρρυθμίσεις που μας χρειάζονται τόσο πολύ για να καταστήσουμε την οικονομία μας πιο αποτελεσματική και πιο βιώσιμη με ανάπτυξη και απασχόληση. Είναι εδώ μια ευκαιρία έχουμε για να υποφεληθούμε ως το δυνατόν περισσότερο των δυνατοτήτων που διαθέτουμε. Και θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα το εξής. Είναι ζώτικο να καταφέρουμε η ΕΤΕ να δώσει προτεραιότητα στα, σχέδια, στα βιώσιμα σχέδια. Τα σχέδια δηλαδή που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενεργείας και προγράμματα που δεν δαπανούν, δεν δημιουργούν πολλές εκπομπές διοξιδίου. Επίσης, τις επενδύσεις που τονίζουν την καινοτομία, την έρευνα, την ανάπτυξη και όπου η χρηματοδότηση τονίζει ιδιαίτερα την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ενεργειακών με λιγότερες εκπομπές διοξιδίου. Επίσης να ενδυναμωθούν τα σχέδια που βρίσκονται ακόμη σε πειραματικό μεν στάδιο αλλά που ακόμη δεν είναι εμπορικά βιώσιμα δηλαδή μια ευρωπαϊκή στρατηγική που να τονίζει περισσότερο τις επενδύσεις και με περιβαλλοντολογική αξιολόγηση και κοινωνική αξιολόγηση. Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στη λεγόμενη Επιτροπή, Επενδυτική Επιτροπή, Επιτροπή Επενδύσεων. Δεν πρέπει να τονίσουμε μόνον το χρηματοδοτικό, το δημοσιονομικό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλες τις πτυχές οικονομικές, περιβαλλοντολογικές για να έχουμε μία πιο ολοκληρωμένη άποψη. Οι επενδύσεις πρέπει να να στοχεύουν ιδίως και περιφερειακούς στόχους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία μου. Αν Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ε, αστεία το είπα, αστεία το είπα. Δεν έχει ρουμανική καμπίνα σήμερα. Λοιπόν, ε, χαίρομαι ιδιαίτερα για την εργασία της Κάτελάιν. Δεν ήταν εύκολη η δουλειά της σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Μπόρεσε να ασχοληθεί με ένα τόσο ευαίσθητο και λεπτό θέμα γιατί όλοι μιλάνε για αυτό το νέο θαύμα, το σχέδιο Juncker. Η ποιότητα της εργασίας της είναι πολύ ψηλή και των σκιωδών επίσης. του συγχαίρω και αυτούς. Εγώ είμαι περήφανος για την Ήτρε, αλλά όταν διάβασα αυτή την έκθεση κατάλαβα ότι είμαι περήφανος γιατί με ενδιέφερε ιδιαίτερα το πώς να εξηγήσω προς τα έξω ότι η Ευρώπη χρειάζεται χρήματα κόβοντας τον προϋπολογισμό της έρευνας. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο πράγμα, δεν μπορούσα να το πω αυτό. Μιλάμε για ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας, μιλάμε για την ανάγκη ανταγωνισμού, αντιμετώπισης του ανταγωνισμού από τις ΗΠΑ, την Silicon Valley και άλλα και να λέμε ότι πρέπει να βρούμε εργαλεία για να τα κτλ. Αλλά η πρώτη επιλογή ήταν πάντοτε να περικοπούν τα χρήματα της έρευνας. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν γιατί η βρήκε άλλη πηγή. Συγκεκριμένα είπε από πού να πάρουμε τα λεφτά και καταφέρνει να ενθαρρύνει και άλλα μέλη της Ήτρε να πούν όχι δεν είναι πρώτη μας επιλογή η περικοπή του προϋπολογισμού της έρευνας. υπάρχουν και άλλοι τρόποι και μας το λέει αυτό πού μπορούν να βρεθούν τα χρήματα. Δεύτερον, αυτό ήταν το πρώτο. Δεύτερον, πού να πάνε τα λεφτά στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Από τα αγαπημένα μου θέματα είναι οι πράσινες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι για βιώσιμη ανάπτυξη από την υποστήριξη αυτών. Το λέει και αυτό ρητά. Τρίτον, η έκθεση αυτή επίσης λέει ρητά στα κράτη-μέλη ότι πρέπει να βρούμε εξυπνότερους τρόπους επένδυσης, επενδύσεων. Συγχαίρω λοιπόν ακόμη μια φορά την Κατελάινε και χαίρομαι ιδιαίτερα που τώρα μπορώ να βγω από εδώ και να πω δυνατά ότι είμαι περήφανος γιατί η Ευρώπη δεν περικόπτει τον προϋπολογισμό της ερεύνης. Ευχαριστούμε πολύ κύριε συνάδελφε. Ίσως δεν χρειάζονται τα ρουμανικά αφού τα είπατε τόσο καλά στα εγγλέζικα. Η κυρία Μούντι. And, uh, Ευχαριστώ. Να προσθέσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου στην ε, Κατλίν για αυτά τα οποία ε, πέτυχε. Συγκεκριμένα θα ήθελα να εκφράσω την απόλυτη στήριξή μου για τις ε, τροπολογίες, για την χρηματοδότηση του μέσου αυτού και το ότι φεύγουμε για από, φεύγουμε από την λογική του να απομακρύνουμε χρήματα από την έρευνα. Και επίσης η προώθηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας για τους λόγους που ανέφερε η Κατλίν. Ε, και βεβαίως ε, να δούμε και την ενεργειακή φτώχεια και αυτό είναι ένα ζήτημα κλειδί. Και βεβαίως έχουμε και τον ρόλο των ε, συμβούλων και το πώς θα πρέπει βεβαίως να φτάσουν πιο κοντά στα κράτη-μέλη και στις επενδυτικές ε, πλατφόρμες. Και βεβαίω ε, καλωσορίζω και τις ε, τροπολογίες που αφορούν την εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων στα κράτη-μέλη. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική η προσθέμενη αξία του, του ΕΦΣΑ, και βεβαίως ε, τέλος να συγχαρώ και πάλι την Καθλίνα αλλά και τους υπόλοιπους από τις ε, υπόλοιπες επιτροπές γιατί αυτή η κοινή προσέγγιση είναι πάρα πολύ σημαντική και βεβαίως ε, καλό είναι να υπάρχει και αποτελεσματική αλλαγή μέσω αυτής της διαδικασίας και να επιτύχουμε βεβαίως και τους στόχους μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω λιγότερο χρόνο για να δείξω ακριβώς τη σημασία της ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Πρώτα απ' όλα να πω πως καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια στην τελευταία θητεία, ειδικά όσον αφορά το ερωτηματολόγιο για, την, για τον ορίζοντα 2020 και βεβαίως ε, να δούμε τι γίνεται σε σχέση με την ανταγωνιστικότητά μας με ΕΙΠΑ και η Ιαπωνία ειδικά στον τομέα της ενέργειας πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και να απεξαρτηθούμε από κάποια πράγματα. Δεύτερον, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν δίνουμε ακόμη περισσότερη έμφαση σε αυτό το θέμα γιατί αυτή τη στιγμή μια πόλη ή ένα νοικοκυριό ή ένα εργοστάσιο ή οτιδήποτε άλλο το αυτοκίνητο γίνει πιο αποτελεσματικό ε, η εξοικονόμηση αυτή γίνεται επάπειρον και έτσι κερδίζουμε πολύ περισσότερα λεφτά οπότε θα πρέπει να φροντίσουμε η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης να είναι εγγυημένη και να σημειώσουμε πρόοδο ε, σε αυτά τα οποία λέμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα λοιπόν αρκούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κρίστιαν Έλα. Άκουσα κάτι. Κάποιο δισταγμό από τον κύριο Τόιλερ. Πρέπει να ξέρουμε ότι εδώ δεν πρόκειται για μπλόφες. Δεν θέλουμε να βγάλουμε χρήματα από το προϋπολογισμό για να τα ξαναβάλουμε στο ίδιο μέρος. Γιατί αυτό θα ήταν μια γρήγορη αλλά άχρηστη λύση και το δισταγμό τον βλέπω στην ερώτηση του αν όλα αυτά δεν είναι παρά μόνο ένας τρόπος κάλυψης και τίποτα συγκεκριμένο. Δέστε το ορίζον το ίδιο, το οποίο χρηματοδοτείται από τα προγράμματα που δεν δουλεύουν. Βάζουν χρήματα από αυτά στο Horizon δηλαδή. Τι Βλέπετε πρακτικά ότι η Κομισιόν με μικροδιαχείριση βρίσκει χρήματα. Το πρόβλημα δεν είναι να αλλάξει ή να μην αλλάξει το MFF. Αυτά είναι θέματα εύκολης λύσης. Κατ' εμένα είναι πολύ σοβαρό να πούμε ότι βρίσκοντας άλλους πόρους ανεξαρτήτως MFF ως front loading. Να δούμε δηλαδή από πού μπορεί να προέρθουν μερικά χρήματα και μετά θα έρθει η αναγκαία αναθεώρηση του πολιετούς Άμα βρούμε άλλες πηγές, λένε, δεν χρειάζεται να ξανανοίξει το πολιτικό, Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Είναι το θέμα της μικροδιαχείρισης και η αδυναμία της πρότασης της Κομισιόν είναι ότι θεωρούν ότι πρέπει να πάρουν χρήματα για την ανάπτυξη και να τα δώσουν σε αναπτυξιακά προγράμματα. Μην ανησυχείτε. Ακόμα και η τωρινή διαχείριση και κατανομή των χρημάτων στον προϋπολογισμό ε, γίνεται με τον τρόπο ακριβώς που προτείνεται. Με τη μικροδιαχείριση υπάρχει λύση. Δεν είναι ότι αρνούμαστε τα πάντα. Όχι. Υπάρχει εδώ δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Κανένας άλλος σκιώδης γιατί στο τέλος θα ξαναπάρει το λόγο η κυρία Βαν Σκιώδη, Σκιώδης, σκιώδης, όχι. Εξ ονόματος της Κομισιόν ο κύριος Ρουγκό. Δεν έχω σχόλιο. Θα τα πείτε με τον Επίτροπο Κατάινεν αύριο. Μια στιγμή, μια στιγμή. Μια στιγμή. Η συνάδελφός μου θέλει να μιλήσει. Ευχαριστώ. Μερικά σχόλια διότι. Να κάνω κι εγώ γιατί το μέσο είναι κατά βάση μία εγγύηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα πρέπει άρα να υπάρχει σχετική γραμμή στον προπολογισμό. Γι' αυτό κάναμε μία πρόταση να χρησιμοποιήσουμε τον ορίζοντα 20, 20 για να εξοικονομήσουμε λεφτά. Αλλά δεν έχουν χαθεί τα λεφτά ε, για την έρευνα, χρησιμοποιούνται διαφορετικά από ε, λεφτά από κονδύλια επιχορήγησης πήγαν σε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο. Παραδείγματο χάρη για τον ορίζοντα 2020 μιλάμε για 3,5% του συνολικού φακέλου για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συνάδελφοι, συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Συνεχίστε, συνεχίστε. Σας ευχαριστώ για την πολύ έντονη συζήτηση και τις απόψεις σας για το πώς ε, πρέπει να διαθέσουμε τα κονδύλια. Θέλαμε η πρόταση να είναι ως το δυνατόν πιο ευέλικτη για να προωθήσει ακριβώς ε, γρήγορα την ε, ανάπτυξη και τις δουλειές στην Ευρώπη. Γι' αυτό δεν προτείναμε ποσόστοση για κάποιο συγκεκριμένο τύπο έργου. Ευχαριστώ. Αυτά ήταν τα βασικά ε, που ήθελα να πω αυτή τη ε, στιγμή. Ευχαριστώ. Θα το συζητήσουμε οπωσδήποτε. Είναι η κυρία Βαμπρέμπτ σε λίγο. Αύριο στις 5.30 και για δύο ώρες με τον κύριο Κατάινεν και τον κύριο Μόρε τους επιτρόπους και οπωσδήποτε όλα αυτά θα απαντηθούν αύριο. νομίζω και από εκεί πέρα είναι σαφής η απόψη. Παρακαλώ να ε, έρθετε και τώρα η συγγήτριά μας. Ε, μα τα αντέξατε τόσα κοπλιμέντα. Κοιτάξτε υπάρχει μια παροιμία στα Ολλανδικά. Θα προσπαθήσω να την ε, μεταφράσω. Δεν ξέρω τώρα αν μεταφράζεται καν. Στα Ολλανδικά λένε πρόσεχε άμα σου δίνουν πάρα πολλά λουλούδια γιατί σε λίγο ακολουθεί και η γλάστρα. Ήταν χτες και η Διεθνής ημέρα των γυναικών, λέει ο Πρόεδρος, οπότε είμαστε μέσα στο κλίμα. Ενθαρρυντικό βεβαίω, ενθαρρυντικά όλα αυτά και όπως είπα αυτό είναι η δουλειά όχι μόνο της ε, εισηγήτριας ε, και των ε, βοηθών μου αλλά και των σκιωδών και είναι το ισχυρότερο μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε και θέλω να πω κάτι για την Κομισιόν οι άνθρωποι είναι υπάλληλοι δεν μπορούν σήμερα να τοποθετηθούν πολιτικά το αντιλαμβάνομαι Αύριο έχουμε δύο επιτρόπους, ο ένας ε, ο υπεύθυνος για την έρευνα και την ανάπτυξη και ο άλλος για την πολιτική της ενέργειας. Οπότε θα τα πούμε μαζί τους. Αλλά οι εκπρόσωποι της Κομισιόν που είναι εδώ πέρα σήμερα, σήμερα σημειώστε παρακαλώ πως θα επιμείνουμε σε αυτές τις θέσεις και προετοιμαστείτε να έχετε κάποιες καλές λύσεις και να συνεργαστείτε μαζί μας, γιατί τελικά πρόκειται για κάτι το οποίο θα βοηθήσει και την Κομισιόν. Γνωρίζω εντό τη γενική διεύθυνση έρευνα και ανάπτυξη Ενέργειας ε, και, τα λοιπά και δεν ξέρω καν αν λέω και σωστά τα ονόματα των Γενικών Διευθύνσεων. Ξέρω πως και εκείνοι πραγματικά κλαίνε όταν πρέπει να κόψουν από τον ορίζοντα 2020 και τον μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Εγώ δεν ήμουν τόσο δραστήρια όσο ο κύριος Έλερ και η Λυπή, αλλά παρακολούθησα το πολιτισμό νομικό πλαίσιο πάρα πολύ στενά και οι προτάσεις που έγιναν της Κομισιόν ε, ήταν πάρα πολύ κοντά σε αυτά τα οποία έλεγε το ε, Κοινοβούλιο παρά το Συμβούλιο. Καταλαβαίνω ότι εσείς είστε υπάλληλοι, αλλά μεταφέρετε τα. Πρέπει να συνεργαστούμε, έχουμε ένα καλό σχέδιο επενδύσεων και όπως είπα, όλοι σχεδόν σήμερα είπαν πως θα ε, υποστηρίξουμε αυτό το σχέδιο σχεδόν, σχεδόν όλοι, εντάξει. Και ακόμα στηρίξαμε και το βασικό ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο προπολογισμό τη Ένωση για εγγυήσει και πρέπει να υπάρχει πράγματι κάποιο αποθεματικό. Αλλά όχι από δύο μεγάλα προγράμματα που ήδη υφίστανται. Οπότε δεν θα το συζητήσω περισσότερο και προτείνω να μην μπούμε στις ε, λεπτομέρειες γιατί αυτό θα το κάνει η διαδικασία του προϋπολογισμού. Εμείς ορίζουμε τις αρχές ότι θα υπάρχει ένα αποθεματικό και μετά επαφίεται στους ε, αρμοδίους ε, του προϋπολογισμού να φροντίσουν να υπάρχουν τα σχετικά κονδύλια για να λειτουργήσει το πρόγραμμα αλλά και βεβαίως να λειτουργήσει και με τα σωστά περιθώρια. Για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα λοιπόν βλέπω κάποιες διαφορετικές ε, προτεραιότητες ε, να εξηγήσω λίγο κάτι. Ότι τώρα δηλαδή υπάρχει ε, αυτό το εύση και θα έχει μόνο προτεραιότητα την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Όχι, θα το διευρύνουμε στο πλαίσιο των γενικότερων όμως γραμμών που έχουμε θέσει στο κλίμα, στην ενέργεια, στον ορίζοντα 2020 κτλ. Να φροντίσουμε λοιπόν οι επενδύσεις που θα κάνουμε να είναι σε αυτό το πλαίσιο. Και ναι, έκανα κάποιες παρατηρήσεις για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα γιατί θεωρώ πως έτσι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας και θα έχουμε τεράστιες επενδύσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον κόσμο που αντιμετωπίζει δυσκολία. Φρόντισα λοιπόν να υπάρχει ένα ευρύ φάσμα. Και τέλος, επειδή ε, δεν το ανέφερα στην ε, εισαγωγή μου, αναφέρθηκα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Ε, εγώ κρίνω με βάση το βέλιο έτσι. Δηλαδή, μια εταιρεία 3.000 ε, υπαλλήλων δεν είναι μικρή πλέον, είναι μεγάλη. Έτσι. Και βεβαίω ε, δικαιούνται και αυτοί στο ΕΨΙ να μπουν αν έχουν σωστά έργα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι το φάσμα, δηλαδή το τι ε, εννοούμε όταν λέμε μικρόμεσαίες επιχειρήσεις. Και για καινοτόμες επιχειρήσεις ε, μεσαίας ε, κεφαλοποίησης. Ε, ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα λουλούδια, τα μεταφορικά. Είναι το πρώτο βήμα και ακόμα και αν καταλήξουμε σε μια πάρα πολύ καλή πλειοψηφία στην Ήτρα, ο πραγματικός αγώνας και οι συζητήσεις θα ακολουθήσουν μετά, όταν θα διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο. Οπότε πρέπει να είμαστε αρκετά ενωμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω και εγώ στη γλώσσα μου. Είδατε ότι φορούσα ακουστικά και άκουσα τη διερμηνία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πολωνική καμπίνα. Θα δούμε λοιπόν τις τροπολογίες αύριο το απόγευμα από τις 5.30 θα έχουμε πάλι συνεδρίαση και θα έρθει να μας μιλήσει στην Ολομέλεια ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Θέλουμε όλοι απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα. Από πού θα βρούμε τα λεφτά για αυτό το πολύ σημαντικό ταμείο. Θα ξαναειδωθούμε λοιπόν αύριο. Σας κατευχαριστώ.